<clears throat> Επαναλαμβάνεται η συνεδρία. Καλημέρα σα, και κύριοι. Το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι έκθεση Wolf Klintz με θέμα του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων όσον αφορά ορισμένου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Ο κύριος Κλίντς, εισηγητής, έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.